πλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την 1η Φεβρουαρίου να καλωσορίσουμε τους νέους συναδέλφους και να τους θυμίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούν τον κανονισμό στις συνεδριάσεις ε, ε, του Κοινοβουλίου και των οργάνων του. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα ε, της ημερήσιας διάταξης που είναι η συνεχιζόμενη απειλή για το κράτος, ε, συγγνώμη, το παράνομο εμπόριο ζώνη συντροφιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προφορική ερώτηση. Έχουμε ε, τους αγορητές, έχουμε τις ε, μπλε κάρτες ε, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης για αυτή τη συζήτηση. Ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση με τον εισηγητή, τον συνάδελφο κύριο Πόλτσακ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που ε, θα συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι ευτυχώς πολύ πιο συνενετικό από το προηγούμενο. Υπάρχει διακομματική συμφωνία για αυτή την προφορική ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το λαθρεμπόριο ζών συντροφιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ρενάτα Ζόμερ κίνησε το θέμα αυτό στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη έχει εκπονήσει πολλαπλά ψηφίσματα για το θέμα αυτό. Αλλά τα λόγια και τα κείμενα δεν αρκούν. Χρειαζόμαστε έργα, συγκεκριμένες πράξεις. Γι' αυτό και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τα κράτη-μέλη, να θεσπίσουν το συντομότερο κάποια μέτρα και να αντιδράσουν αποτελεσματικά. Γιατί μας ενδιαφέρει η καλή μεταχείριση των ζώων, μας ενδιαφέρει η ευζόεια και εδώ μιλούμε για εκατομμύρια καταναλωτές, ε, συμπολίτες μας ε, που επηρεάζονται πολύ αρνητικά από το λαθρεμπόριο αυτό. Γιατί το λαθρεμπόριο δεν γνωρίζει σύνορα και το λαθρεμπόριο των ζώων συντροφιάς αποφέρει τεράστια κέρδη. Είναι η τρίτη πιο επικερδής ε, παράνομη δραστηριότητα μετά το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών το λαθρεμπόριο των ζώων συντροφιάς. Επίσης, ε, έχουμε εκτροφή γάτων και σκύλων σε άθλιες συνθήκες με μοναδικό στόχο το λαθρεμπόριο του στη συνέχεια για την αποκόμιση κέρδους. Εμείς ε, θέλουμε καλή μεταχείριση των ζώων και πολλές φορές ε, εκδίδονται πλαστά έγγραφα για τα ζώα αυτά, πλαστά διαβατήρια, πλαστά πιστοποιητικά σωστής εκτροφής και ε, πολύ συχνά εξαπατώνται οι πολίτες να αγοράσουν αυτά τα κουταβάκια και τα γατάκια που έχουν εκτραφεί σε πραγματικά άθλιες και παράνομες συνθήκες. Και ακριβώς επειδή είναι χαμηλό το τίμημα πώληση, ε, πολλοί καταναλωτές πέφτουν στην παγίδα και αγοράζουν τέτοια ζώα που είναι θύματα αυτού του λαθρεμπορίου των ζώων συντροφιά. Και οι λαθρέμποροι βρίσκουν τρόπους και παραθυράκια για να παρακάψουν την ε, κοινοτική νομοθεσία. Πολλά ε, κουτάβια που εκτρέφονται με αυτόν τον τρόπο είναι άρρωστα. Είναι λόγω της, ε, των κακών συνθηκών εκτροφής έχουν κακή υγεία. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε και μία ε, ζωνόσο, μία επιζωοτία λόγω αυτών των κακών συνθηκών εκτροφής. Και μάλιστα είχαμε και μόλις 30 ανθρώπων. Αυτό το λαθρεμπόριο λοιπόν ζώων συντροφιά έχει πολύ αρνητικέ συνέπειες ε, και στην εσωτερική αγορά και στην προστασία των, του καταναλωτή, γιατί πολύ συχνά οι καταναλωτές αγοράζουν είτε άρρωστα ζώα, είτε ζώα που είναι τραυματισμένα λόγω των άθλιων συνθήκων εκτροφής τους. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης, να καταπολεμήσει την παραπληροφόρηση και να ρυθμίσει τις επιγραμμικές πωλήσει ε, γατιών και σκυλιών. Επίσης, ε, η απάνθρωπη μεταχείριση των ζώων είναι μια μάστιγα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή λύση γιατί πρόκειται για ένα διασυνοριακό πρόβλημα. Θέλουμε έναν πανευρωπαϊκό τρόπο εντοπισμού, ταυτοποίηση και εγγραφή των ζώων συντροφιά. Θέλουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα ταυτοποίηση των ζώων συντροφιάς ώστε να ταυτοποιούνται όχι μόνο τα ζώα συντροφιά, αλλά και τα δέσποτα ζώα και να καταπολεμήσουμε την κακή τους μεταχείριση σε παράνομες μονάδες εκτροφής Έχουμε κάθε χρόνο θύματα εκατομμύρια κουταβάκια και γατάκια. Θέλουμε λοιπόν καλύτερες επιθεωρήσεις και ελέγχους, πιο συχνούς κτηνιατρικούς ελέγχους και οι κτηνίατροι πολλές φορές ελέγχουν μόνο νόμιμες μονάδες εκτροφής και οι παράνομες τέτοιες μονάδες εκφεύγουν του κτηνιατρικού ή οποιοδήποτε άλλο ελέγχο. Περιμένουμε λοιπόν προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά αυτή τη μάστιγα που είναι το λαθρεμπόριο των ζώων συντροφιά. Γι' αυτό απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να μεριμνήσουν για να απαλλαγούμε αυτή τη μάστιγα και να προστατεύσουμε ανθρώπους που είναι ανήμποροι και δεν μπορούν να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Νικολίνα Μπρνιάτς από το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Τα πρόσφατα χρόνια το παράνομο εμπόριο ζών συντροφιάς αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ανησυχίες ε, στους πολίτες, ιδιαίτερα ως προς την ανάπτυξη των ε, επιγραμμικών πωλήσεων των ζώων συντροφιάς και τους ε, συναφείς ε, κινδύνους. Ξέρετε ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, όχι μόνο ως προς τη δημόσια υγεία και την προστασία των καταναλωτών, αλλά και για την υγεία των ζώων. Θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη προσοχή σε αυτό το ζήτημα. Το γνωρίζουν τα κράτη-μέλη. Τα τέλη του 2018-17 κράτη-μέλη συμμετείχαν σε ένα συντονισμένο ε, σχέδιο ως προς τις επιγραμμικές ε, πωλήσει ζώων συντροφιάς και δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό πωλήσεων ε, δεν συμμορφούτο προς τους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την ευθύνη που φέρουμε και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβάλλει κανόνες ως προς την ε, εισαγωγή αυτών των ζώων. Επίσης υπάρχει ένα αριθμιστικό πλαίσιο ελέγχων για να μην υπάρχει παράνομο εμπόριο. Χρειάζεται η σωστή εφαρμογή των κανόνων και ρυθμίσεων. Αυτό αποτελεί ευθύνη της Επιτροπής και των κρατών μελών. Από την, μετά από την έγκριση του νέου κανονισμού για τους κτηνιατρικούς ελέγχους των ζώων προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε το παράνομο εμπόριο στα ζώα συντροφιάς. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία όλων των αρμοδίων αρχών μεταξύ των κρατών μελών. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις στην ομάδα εργασίας ως προς το ηλεκτρονικό εμπόριο και την νέα πλατφόρμα σε σχέση με τις επιγραμμικές πωλήσει και εμπόριο. Το Συμβούλιο στα πρόσφατα συμπεράσματά του για την ευημερία των ζώων ενθάρρυνε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τη νομοθεσία για την ευημερία των ζώων. Επίσης, θα δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ερχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επίτροπος, ε, η κυρία Κυριακίδη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Πρόκειται για ένα θέμα για το οποίο προσωπικά έχω πολύ δυνατά αισθήματα. Εμείς ε, ε, πραγματικά ε, πρέπει, είμαστε, έχουμε δεσμευτεί να ελέγξουμε και να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο. Όμως κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίζει το γεγονός ότι τα ζώα συντροφιάς και το καθεστώς τους ε, ε, είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών ε, που έχουν την αρμοδιότητα για την ευημερία αλλά και για την ταυτοποίηση, την καταγραφή και την κίνηση των ζώων αυτών στο εθνικό τους στην εθνική τους ε, επικράτεια. Ε, υπάρχουν ε, ξεκάθαροι κανόνες βέβαια και για τις εμπορικές και τις μη εμπορικές μετακινήσεις. Τα, οι μετακινήσεις ζώων που εντός της Ευρωπαϊκής και Ένωσης και εκτός αυτής ρυθμίζονται επίσης από κανόνες. Μιλάμε για την ευημερία των ζώων αλλά και για ζωνόσους και ειδικά για την λύσα. Υπάρχουν κατοικίδια όπως ε, σκύλοι και γάτες που μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ταυτοποιούνται και να εμβολιάζονται. Αν δεν ε, ταυτοποιούνται, αυτό δεν συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία, απλώ ε, δεν εφαρμόζεται σωστά από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε περισσότερη ενέργεια σε αυτό το θέμα. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε το νομικό πλαίσιο για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το παράνομο ε, εμπόριο. Ο νέο κανόνα που θα μπει σε ισχύ τον ε, Απρίλιο του 2021 θα ζητά την ε, υποχρεωτική νομοθεσία για όλα τα εγκαταστάσεις που δέχονται σκύλους και γάτες αλλά και για κάθε μετακίνηση αυτών των ζώων. Δεύτερον, θα υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τα καταφύγια και γενικά συνθήκες μετακίνησης ε, των ζώων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Επίσης ε, θα ελέγξει καλύτερα το εμπόριο των ζώων συντροφιάς και θα έχει τα απαλκή μέτρα για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου. Είναι κρίσιμο όμως, να εφαρμοστούν σωστά αυτοί οι κανόνες και γι' αυτό έχουμε αναλάβει δράση σε διάφορα κράτη-μέλη. Πρώτον, έχουμε ένα συντομισμένο πλαίσιο για το, την ασφαλή πώληση ε, ζώων σκύλων και γατών. Επίσης ε, θέλουμε να ελέγξουμε το επιγραμμικό εμπόριο αυτών των ζώων. Υπάρχει επίσης ε, και η πρωτοβουλία, θελοντική πρωτοβουλία, η οποία είναι της υπομάδας για την υγεία και την Ευημερία των ζώων συντροφιάς και υπάρχει και η πλατφόρμα για την Ευημερία των ζώων αυτά ε, ε, συνοδεύονται από την καλύτερη εκπαίδευση των εθνικών αρχών που ενισχύουν ε, τις βέλτιστες πρακτικές στην εισαγωγή και το εμπόριο σκύλων και γατών. Επίσης υπάρχει και μια εξέλιξη ως προς την διασύνδεση των βάζων δεδομένων. Βέβαια είναι θέμα αναλογικότητας. Υπάρχει, μια αναλογη... υπάρχει δυσανάλογη επίπτωση στην υγεία των ζώων χωρίς να υπάρχει προστιθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και τα ενδιαφερόμενους ώστε να σταματήσει το παράνομο εμπόριο κατοικιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Ξεκινάμε τον πρώτο γύρο ε, με τον συνάδελφο Μαζίλη από, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό, ε, από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σα Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο στρατηγός Σβάικ ξεκίνησε εκτροφή σκύλων. Τώρα το εμπόριο έχει ξεχρονιστεί, μπορούμε να αγοράσουμε και μέσω του διαδικτύου κουτάβια, αλλά δεν λαμβάνουμε υπόψη τους δυνητικούς κινδύνους. Έχουμε πολλά παραδείγματα μετάδοσης ε, ζωνόσων στους ανθρώπους. Είχαμε ε, το πρόσφατο κορονοϊό και ε, το λαθρεμπόριο κατοικιδίων αυξάνει το κίνδυνο μετάδοση ζωνός, όπως είχαμε πολλά κρούσματα λύσας στις κάτω χώρες. Επίσης, οι ακατάλληλες συνθήκες μεταφοράς οδηγούν σε θάνατο των κατοικιδίων. Τα κατοικίδια, τα ζώα συντροφιά είναι ζωντανά πλάσματα, δεν είναι αντικείμενα, δεν είναι προϊόντα αγοραπολισίας απλώς. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση στο πρόβλημα που είναι διασυνοριακό. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρουμε την έλλειψη επιστημονικής έρευνας στον τομέα αυτό. Επίσης, θα πρέπει να επιβάλλουμε αυστηρότερες κυρώσεις κατά των λαθρεμπόρων κατοικιδίων ζώων. Σας ευχαριστώ κυρία Σπούρεκ, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, παρακαλώ δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάθε χρόνο ε, μεγάλος αριθμός ζώων συντροφιάς είναι αντικείμενο λαθρεμπορίου στα κράτη-μέλη. Πολύ συχνά υποβάλλονται τα ζώα αυτά σε μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων χωρίς τροφή και νερό. Και μάλιστα οι αρνητικές συνέπειες αυτού του λαθρεμπορίου δεν αφορούν μόνο τα ίδια τα ζώα, αλλά και την δημόσια υγεία και την προστασία του καταναλωτή. Θα πρέπει να επιβάλλουμε λοιπόν αυστηρές κυρώσεις κατά των λαθρεμπόρων, καλύτερη αστυνομική συνεργασία, καλύτερη δικαστική συνεργασία και αυστηρότερες προδιαγραφές υγείας των ζώων. Θέλουμε κατάρτιση των διοκτικών μέσων και των αστυνομικών, ώστε να εντοπίζουν καλύτερα περιπτώσεις τέτοιου λαθρεμπορίου κατοικιδίων. Θέλουμε αυστηρότερου κανόνε για την ταυτοποίηση και την καταγραφή επίσης γάτων και σκυλιών, καθώς και την καταγραφή και την αδειοδότηση όλων των εκτροφέων και πολιτών ζώων συντροφιά. Τα συστήματα επίσης καταγραφής θα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένα μεταξύ των κρατών μελών και γιατί 8% του λαθρεμπορίου κατοικιδίων γίνεται μέσω του διαδικτύου. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και αυτή τη διάσταση και περισσότερες εξαιρετικές επιστοπίσεις για να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις αρνητικές συνέπειες του λαθρεμπορίου ζώων συντροφιά και να επισημάνουμε τη σημασία που έχει η αγορά ζώων συντροφιά που έχουν εκτραφεί και ε, ε, πολιθεί με τρόπο που σέβεται την ευζοία και την καλή τους μεταχείριση. Θέλουμε περισσότερη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για να ενθαρρύνουμε την υιοθεσία και όχι την αγορά τροφιάς. Αν περισσότεροι συμπολίτε μας υιοθετούν κατοικίδια αντί να αγοράζουν και έχουμε καλύτερη έρευνα των εκτροφέων, θα χτυπήσουμε έμεσα τους λαθρεμπόρους και έτσι σιγά σιγά θα εξαλειφθεί αυτή η μάστιγα. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Renew Europe το λόγο έχει ο κύριος Χόισικ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, 100.000 κουτάβια. Αυτό είναι η εκτίμηση του αριθμού των ε, κουταβιών που κάθε χρόνο εξάγονται από τη χώρα μου την Σλοβακία και είναι εκτίμηση γιατί ένα μεγάλο κομμάτι αυτού είναι παράνομο εμπόριο. Το εμπόριο δεν είναι πρόβλημα μόνο για την ευμερία των κουταβιών ε, και των ε, ε, άλλων μικρών ζώων. Είναι ένα πρόβλημα γιατί συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα, μέσα στα πλαίσια της κινητοποίησης για την ευμερία των ζώων είδα ακριβώς πώς συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, πώς δίνονται τα χρήματα για την αγορά όπλων. Επίσης, είναι θέμα απώλειας φορολογικών εσόδων, αλλά και θέμα ανθρώπινων ανθρώπινης υγείας. Υπάρχει ένα νέο φαινόμενο που έχει κυριαρχήσει σε όλο το εμπόριο. Είναι οι online πλατφόρμες. Αυτό αυτές ε, έχουν κάνει το πρόβλημα ακόμα πιο ευρωπαϊκό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της και να δώσει την κατάλληλη καθοδήγηση για να γίνεται σωστή ταυτοποίηση και καταχώρηση των ζώων ε, και εκτός συνόρων, αλλά και τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει να ξεκινήσουν να εφαρμόζουν σωστά τους κανονισμούς, ειδικά για την ευζοία των ζώων. Γιατί αυτό που αντιμετωπίζουμε στη φάση αυτή είναι μια κρίση και το μόνο που χρειάζεται είναι δράση, όχι λέξεις και λόγια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον συνάδελφο Ντρεώστο από την ομάδα ID. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, η, παράνομη εμπορία των ζώων συντροφιάς δεν θα πρέπει να γεμίζει ορισμένες ε, τσέπες. Δυστυχώς υπάρχουν στην Ιταλία 400.000 ζώα συντροφιάς και ιδιαίτερα στην περιοχή Φριούλη Βενέτσια Τζούλια εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο ε, από ζώα συντροφιά, τα οποία προέρχονταν από την πρώην Ανατολική Ευρώπη τα οποία μεταφέρονταν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε αυτό το παράνομο εμπόριο των ε, μικρών ζώων συντροφιάς. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασυνοριακή συνεργασία, ιδιαίτερα των ε, τελωνιακών αρχών που πλήττουν τα μικρά και συμπαθητικά τετράποδα. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τον συνάλφα Γκερέρο εκ μέρου ε, των Πράσινων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι ένα ε, bulldog φτάνει από 350 ευρώ μέχρι τα 1600 ανάλογα από τη χώρα. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η μαύρη αγορά, διότι μεταφέρονται αυτά τα ζώα εκεί όπου μπορούν να αποδώσουν περισσότερο. Επίσης δεν υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Μητρό εκτροφέων. εκτροφέων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ζώα αυτά μεταφέρονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει νομοθεσία που να επιβάλλει επίσημα μητρό όλων των ζώων συντροφιάς έτσι ώστε να υπάρχει και διασταύρωση στοιχείων και μητρών. Δυστυχώς όμως πιστεύω ότι χωρίς αυτά τα μητρώα θα αποτύχουμε. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε με τη συνάδελφα Χάζεκαμπ από την ε, Γκουε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τα κατοικίδια ζώα προσφέρουν πολλές χαρές, αλλά δυστυχώς ε, ε, το εμπόριο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και οδύνες τα ζώα. Οι συνθήκες εκτροφής και μεταφοράς είναι άθλιες. Ε, πολλά ζώα είτε είναι αντικείμενα κακής μεταχείρισης ή και ακόμη και θανάτου γνωρίζετε ότι ε, τα ισπανικά κυνηγός και τα τιμωρούν μερικές φορές ε, ε, και από την εξάντληση πεθαίνουν ή μερικές φορές βρίσκονται ακόμη και κρεμασμένα. Επίσης έχουμε πολλές περιπτώσεις κακής μεταχείρισης των ζώων ε, δηλητηριασμούς, πυροβολισμούς, ε, τους κόβουν την ουρά, τα αυτιά, πνίγουν τα ζώα. Και επίσης με το λαθρεμπόριο κουταβιών, η εκτροφή γίνεται μαζικά σε τεράστιες αποθήκες και η πώλησή τους μέσω του διαδικτύου. Θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτό το λαθρεμπόριο, να γίνει υποχρεωτική η καταγραφή των ε, ζώων αυτών, γατιών και σκυλιών να έχουν μια ηλεκτρονική ταυτοποίηση και να χτυπήσουμε το οργανωμένο έγκλημα και τα δεινά των καημένων αυτών κατοικιδίων. Η κυρία Εύη από τους μη εγγεγραμμένους. Όποιος αγοράζει ένα ε, σκυλάκι ε, δεν ξέρει ότι ενισχύει το οργανωμένο έγκλημα είναι το πιο προσοδοφόρο επάγγελμα μετά από την πώληση όπλων και ναρκωτικών. Δυστυχώς αυτά τα μικρά ζώα είναι πολύ ευάλωτα, μεταφέρονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες και μόνο το ίμιση αυτών επιβιώνει αυτή της απάνθρωπης μεταφοράς. Αυτός ο εφιάλτης θα πρέπει να σταματήσει. Θα πρέπει να υπάρχει ε, μία υποχρεωτική καταγραφή και μητρώα, δηλαδή τράπεζες δεδομένων που να ε, συνδέονται μεταξύ τους για να υπάρχει η, η χνηλάτιση των ζώων. Επίσης ένα κυρωτικό πλαίσιο που να αφορά και εκτινιάτρους που πολλές φορές συνεργάζονται. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο αριθμό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, εκπρόσωπε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, εμείς ε, θεωρούμε ότι τα σκυλιά και τα γατιά είναι φωσιωμένοι μας φίλοι. Αν ε, έχει μεγαλώσει κανείς σε μια φάρμα, πάντοτε έχει κοντά του τέτοια ζώα. Πολλοί όμως σκύλοι και γάτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τυχάνουν χάνουν σωστής μεταχείρισης. Μάλιστα, το παράνομο εμπόριο και υπάρχουν ε, αντίξωες συνθήκες εκτροφής. Ε, μάλιστα, ε, δεν δίνεται κτηνιατρική φροντίδα για να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος. Προτείνω λοιπόν αφενός να υπάρχουν πιο αυστηροί έλεγχοι στα κράτη-μέλη, γιατί είναι η αυτό των κρατών μελών, όχι της Κομισιόν, το ξέρω, αλλά χρειάζεται να υπάρχουν ενιαία στάνταρ, ένα ενιαίο σύστημα καταχώρησης που να συνδέεται με βάσεις δεδομένων και να υπάρχει καλή καλύτερη ρύθμιση του, συμβουλ... του εμπορίου στο ίντερνετ. Στην Βαλονία που προέρχομαι υπάρχει μια καλή ρύθμιση του εμπορίου ε, στο διαδίκτυο και έτσι διασφαλίζεται καλύτερες συνθήκες. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον συνάδελφο Τσιου Τσοχαντάρου. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώντας ε, για αυτό το σημαντικό ζήτημα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ε, και ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα. Εγώ έχω συνεργαστεί στο Ιάσιο, σε, στο τοπικό νοσοκομείο και σε μία κτηνιατρική κλινική. Στην ε, χώρα μου δυστυχώς βασανίζονται τα ζώα. Και ευτυχώς υπάρχουν κυρώσεις μέχρι και φυλάκιση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις μολυσματικές ασθένειες των ζώων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως βλέπουμε ότι ισχύει και τώρα, όχι μόνο σε επίπεδο ζωονόσων, γενικών ζωονόσων, αλλά και σε επίπεδο κορονοϊού. Γι' αυτό χρειάζεται ε, ε, εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των ζώων. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον συνάδελφο Χόιτεμα. Yes. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε. Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Μου έκαναν δώρο ένα κουταβάκι και ίσως ήταν το ομορφότερο δώρο που έλαβα ποτέ. Και μάλιστα αυτό το κουταβάκι συνέχισε ε, να περνάει τη ζωή του στη αγροτική μας εκμετάλλευση. Δυστυχώς δεν είναι χαρισάμενη έτσι η ζωή όλων των κατοικιδίων. Πολύ συχνά η εκτροφή τους γίνεται σε ανθυγιεινές συνθήκες, με κακή μεταχείριση, δεν βλέπουν το φως της ημέρας και πολύ συχνά αγοράζονται καλόπιστα από κάποιους καταναλωτές. Τα ζώα μας αυτά είναι ήδη άρρωστα και τραυματισμένα και ψυχικά, κάτι που επηρεάζει και την συνέχεια της ζωής τους. Ο αγοραστής θα πρέπει να βρει κτηνίατρο για να τα φροντίσει, η συντήρησή τους γίνεται δαπανηρή η κατάσταση είναι απαράδεκτη λοιπόν και θα πρέπει να καταπολεμηθεί αυτό το λαθρεμπόριο των κατοικιδίων. Η κυρία Μέτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάθε χρόνο χιλιάδες ζώα συντροφιάς είναι το αντικείμενο λαθρεμπορίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ζώα αυτά πολύ νωρίς τα χωρίζουν από τη μητέρα τους, δεν τρέφονται σωστά, είναι άρρωστα, ε, ε, τη κακής μεταχείρισης και ε, πολλούνται παρά, παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, γιατί είναι φορεί λιμωδών νόσων και οι καταναλωτές πολύ συχνά αγοράζουν αρρωστημένα ζώα, τραυματισμένα και χρειάζεται να ξοδέψουν πολλά χρήματα στους κτηνιάτρους θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει την εχνηλασιμότητα, προτείνοντα ένα εναρμονισμένο σύστημα καταγραφή αυτών των ζώων και επίση να σταματήσουν οι επιγραμμικέ παράνομε διαφημίσει. Θα πρέπει να απαιτούμε συστηματική ταυτοποίηση των πολιτών. Επίσης θα πρέπει να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη για να εξαρθρωθούν τα κυκλώματα των λαθρεμπόρων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε όλα αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα λαθρεμπορίου. Ευχαριστώ κύριο Σκομίνη Ολιβέρες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κανονισμός 567 ε, του 2013 αναφερόταν σε μη εμπορικές διακινήσεις ε, των ε, ζώων συντροφιάς. Το λαθρεμπόριο των κατοικιδίων παραβιάζει το κανονισμό και επίσης επηρεάζει και την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Γιατί μιλούμε πολύ συχνά για διαδικτυακό εμπόριο. Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι σαφές για την ε, λύση του προβλήματος. Θα πρέπει να εφαρμόζεται καλύτερο ο κανονισμός, να επιβάλλονται κυρώσεις ε, στους δράστες και σε πολιτές, ε, διαφημιστές, κτηνιάτρους, θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα καταγραφής και ταυτοποίησης γατιών και σκυλιών και ευαισθητοποίηση των πολιτών προκειμένου να υιοθετούν και να μην αγοράζουν ζώα συντροφιά και καλύτερη συνεργασία των αστυνομικών και τελωνιακών αρχών. Αυτό είναι ο δρόμο. Και α μην ξεχνούμε ότι η ευζοία έχει άμεση σχέση με την ευημερία των ανθρώπων. Γιατί το λαθρεμπόριο ζώων που δεν είναι εμβολιασμένοι, δεν έχουν τα είναι, δημιουργεί ένα πρόσφορο έδαφο για τη μετάδοση κενώσεων. Θέλουμε μια κοινωνία που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. Μια τέτοια κοινωνία είναι και πιο ανθρώπινη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε τη συνάδελφο Γκλάβεκ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κάθε μήνα υπολογίζεται ότι Περίπου 46.000 σκυλιά είναι αντικείμενα αγοραπολισία, χωρίς να είναι καταγεγραμμένα, χωρίς να είναι εμβολιασμένα, χωρίς να έχουν πιστοποιητικά. Και πολλά από τα ζώα αυτά, αμέσως σχεδόν μετά την αγοραπολισία, πεθαίνουν. Και μάλιστα είναι το τρίτο πιο επικερδές λαθρεμπόριο, το λαθρεμπόριο κατοικιδίων, μετά το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Είναι μάστιγα αυτό το λαθρεμπόριο με αρνητικέ συνέπειε και για την ανθρώπινη υγεία, για την ευζοία και την προστασία του καταναλωτή. Γι' αυτό και η ταυτοποίηση και η καταγραφή όλων των αγαθιών και σκυλιών είναι το πρώτο βήμα στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου αυτού. Και μάλιστα από πέρυσι το Δεκέμβριο ε, στη διάρκεια της Φιλανδικής Προεδρίας το Συμβούλιο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση του κατά πόσο χρειάζεται νέα νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων. Στην Κροατία έχουμε πολύ καλές ε, διατάξεις για την ευζοία. Ε, Δυστυχώ, τα στοιχεία που έχουμε για το λαθρεμπόριο δημιουργούν μια θλιβερή εικόνα για την πραγματικότητα που θα πρέπει οπωσδήποτε να την αλλάξουμε. Σα ευχαριστώ. Ωραία, συνεχίζουμε με το ΚΑΤΣΔΙΑ. Έχουμε μόνο δύο τέτοια αιτήματα, οπότε θα τα πάρουμε και τα δύο. Ω, oh, συγγνώμη, λάθος μου. Ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει άλλος ένας ε, ε, στη συζήτηση, είναι η συνάδελφος κυρία Ντινόλφη. Σας ζητώ συγγνώμη, πήγα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Το άρθρο 13 της Συνθήκης της ε, Λισαβόνας τονίζει την ευημερία των ζώων, την οποία θα πρέπει να τηρήσουμε και να σεβαστούμε. Δυστυχώς όμως ε, ε, γίνονται απάνθρωπες μεταφορές κουταβιών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υφίστανται μεγάλη ψυχολογική αλλά και σωματική βία. Ε, δυστυχώς ε, ε, βλέπουμε ότι πολλοί πολίτες δεν μπορούν να ταξιδέψουν με τα αγαπημένα του ζώα. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τις εναέριες μεταφορές. Και γι' αυτό βάζουν αυτά τα ζώα στην άτρακτο και τα χρησιμοποιούμε σαν αντικείμενα. Θα πρέπει λοιπόν ακόμα και οι αεροπορικές εταιρείες να επιβάλλουν τη μεταφορά αυτών των ε, ζώων υπό ανθρώπινες συνθήκες. Ευχαριστώ και άλλη μια φορά συγγνώμη που σας ε, πέρασα. Πάμε τώρα ε, στην διαδικασία Κατσδιάη. Έχω μόνο δύο τέτοια αιτήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, είπατε στην εισαγωγική σας ομιλία ότι το λαθρεμπόριο ζώων συντροφιάς είναι εθνική αρμοδιότητα. Αυτό όμως δεν ισχύει. Γιατί θέλουμε πιο αυστηρές κυρώσεις για την καταπολέμηση του λαθρεμπόριου αυτού και πιο αυστηρές ε, ε, διατάξεις ε, και πρότυπα για τα εκτροφία. Άλλωστε, το λαθρεμπόριο είναι μια εγκληματική δραστηριότητα διασυνοριακού χαρακτήρα που πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες ζώα που είναι τα θύματα και υποφέρουν από αυτή την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει αποτελεσματικά μέτρα δεν μπορούν τα κράτη-μέλη μόνα τους ε, να αναχαιτήσουν τέτοιο διασυνοριακό λαθρεμπόριο. Σας παρακαλώ λοιπόν να μεριμνήσετε για το πρόβλημα αυτό. Γιατί ήσταν πολύ γενικοί και όριστοι στην ε, εισαγωγική σας ομιλία. Μιλούμε για α, λαθρεμπόριο που οδηγεί και σε απόλυτα απόλυτα φορολογικών εσόδων, αλλά και οδύνει σε αθώα πλάσματα όπως είναι τα ζώα. Κύριος Οστρεβίτσιους, σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Ευρώπη μάλλον έχει καταργήσει εδώ και ε, πολλά χρόνια το δουλεμπόριο. Είναι δυνατόν όμως τον 21ο αιώνα να μην έχουμε κατάλληλες ε, συνθήκες εκτροφής και μεταφοράς για τα κατοικίδια, τα ζώα συντροφιάς μας. Έχουμε υψηλά πρότυπα στην οικονομία μας και είμαστε πρωτοπόροι στην καινοτομία και τις τεχνολογίες. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε την πολιτική βούληση να θεσπίσουμε ένα εναρμονισμένο σύστημα καταγραφής και ταυτοποίησης των κατοικιδίων ζώων. Καμαρώνουμε και περηφανευόμαστε για τα επιτεύγματά μας, αλλά δεν έχουμε ακόμη ένα ενιαίο μητρό και μια ενιαία βάση δεδομένων για τα κατοικίδια ζώα. Μιλούμε για λαθρεμπόριο που πειράζει τη δημόσια υγεία και την προστασία του καταναλωτή. Γιατί αν δεν επιβάλλουμε αυστηρέ κυρώσει, είναι σαν να αφήνουμε ελεύθερο το λαθρεμπόριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να λάβει άμεσα δράση για να επιβάλλει την καλή μεταχείριση των ζώων και να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή τη σύγχρονη μορφή δουλεία. Ευχαριστούμε και τώρα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Επίτροπο κυρία Κυριακίδη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις παρεμβάσεις σας. Αυτό που δεν χρειάζεται να κάνετε είναι να με πείσετε ότι χρειάζεται να γίνουν περισσότερα πράγματα. Ε, είμαι και εγώ περήφανη ιδιοκτήτρια ενός οικοστού ε, ζώου, επίσης, ε, ενός ζώου συντροφιάς. Επίσης, τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ το επιγραμμικό εμπόριο και μπορώ να πω και παραδέχομαι ότι πολλά από αυτά που βλέπουμε σύμφωνα με τόσο έχω παρακολουθήσει, είναι λυπηρά, ακόμα και σοκαριστικά. Δεν χρειάζεται να με πείσετε λοιπόν ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Να ξαναπώ λοιπόν ότι η Επιτροπή και εγώ προσωπικά έχουμε δεσμευτεί να βρούμε τρόπους να σταματήσουμε το παράνομο εμπόριο γατιών και σκυλιών. Επίσης ε, θεωρώ ότι ο νέος νόμος ε, για την υγεία των ζώων θα αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Έχουμε ε, συγκεκριμένα νομοθεσία για τα εκτροφία ζώων συντροφιάς. Συγκεκριμένα πρόκειται για πιο πολλά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν από τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παράνομες πρακτικές. Το πιο σημαντικό όμως είναι η εφαρμογή των κανόνων, γιατί κατανοούμε ότι δεν εφαρμόζονται οι κανόνες. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να παίξουν το ρόλο που τους αρμόζει σε αυτή την κατεύθυνση και πρέπει ε, να ξεκινήσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Επίσης, ε, ο κανονισμός ε, της Επιτροπής ε, εφαρμόζει πολύ μεγαλύτερα πρόστιμα και κυρώσεις για να σταματήσει το παράνομο εμπόριο. Γιατί πραγματικά το εμπόριο αυτό είναι μια απειλή για την εσωτερική αγορά, για την υγεία και ζωή των ζώων. Και εγώ ως Επίτροπος δεσμεύομαι ότι θα εξετάσω το θέμα πιο στενά και θα δω πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος για την υγεία των ζώων και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι είναι απαραίτητο. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο και έτσι κλείνει ε, η συζήτηση με την εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Μπρίντσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ε, χρήσιμη συζήτηση για την προστασία της εσωτερικής αγοράς και τα δικαιώματα των καταναλωτών από αυτό το παράνομο, παράνομο εμπόριο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο κρατών μελών έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι κανόνες ε, που έχουν εγκρίνει οι συνομοθέτες. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ευημερία των Ζώων αποτελούν σημαντική συνεισφορά σε αυτό το τομέα και πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ως προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνω λοιπόν τη συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, ε, ε, να πω ότι αύριο θα γίνει η ψηφοφορία για το ψήφισμα ε, που 2019-2018 το οποίο ε, επίσης ε, θα βρείτε και στο στο σελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δείτε και εκεί και τη μερίσια διάταξη. Ε, με αυτό κλείνουμε τη σημερινή μας συνεδρία. Ευχαριστώ.